Ευχαριστώ ιδιαίτερα που βρεθήκατε εδώ σήμερα. Η μερίσια διάταξη προβλέπει τι δηλώσει του Συμβουλίου και τη Επιτροπή, οι προτεραιότητε του Κοινοβουλίου εν ώψη τη Συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Γενέβη, 1 με 26 Μαρτίου 2010. Αρχίζουμε τη συζήτηση εξ του Συμβουλίου. Ας δώσουμε ένα λεπτό περίπου για να γίνει η αλλαγή της φουράς. δύο λεπτά. I'm sorry, Ms. Benova, did you ask for the floor? Κυρία Μπένοβα, στήσατε το λόγο. Όχι. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, επαναλαμβάνω. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τι δηλώσει Συμβουλίου και Επιτροπή, οι προτεραιότητε του Κοινοβουλίου εν ώψη τη Συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, Γενέβη 1 με 26 Μαρτίου 2010. Εξ ονόματος του Συμβουλίου, τον λόγο έχει ο κύριος Λόπες Γκαρίδου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει στη Γενέβη, στις Βρυξέλλες και σε πρωτεύουσες τρίτων χωρών την, ε, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Πρόκειται για ένα φόρουμ όπου εξετάζουμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα μέρη του κόσμου και βλέπουμε ποιες είναι οι διεθνείς προσπάθειες για τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Άλλωστε, ε, αυτό είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά, η πεμπτουσία της Ένωσης, ε, στοιχείο της ε, ψυχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που χαρακτηρίζει και την ταυτότητα της Ένωσης και το πρόσωπό της στον κόσμο. Η Προεδρία του Συμβουλίου παίρνει πολύ σοβαρά υπόψη το ρόλο που έχει να διαδραματίσει αυτή τη στιγμή εν ώψη αυτού του Συμβουλίου και λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Γι' αυτό και θα δώσουμε το παρόν ε, με την, αντιπρόεδρο του... της ε, Ισπανικής Κυβέρνησης, τη Μαρία Τερέζα Φρανταγκράβεγκα, ως Προεδρεύουσα του Συμβουλίου και θα ε, κηρύξει την έναρξη τη 13η ε, Συνόδου Εργασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ω εκ τούτου, η Ισπανική Προεδρία θα έχει πολύ δραστήριο ρόλο και παρουσία στι εργασίε του Συμβουλίου. Θα προσπίσουμε τι θέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα που έχουν ε, άμεση συνέπειε για πολλές χώρε μέλη. Και πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποβάλει και ψηφίσματα ειδικά. Πιστεύουμε ότι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χρειάζεται μηχανισμούς για να μπορέσει να προασπίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, για να αντιμετωπίσει κατάφορες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είτε μέσω μιας εντολής για συγκεκριμένη χώρα, όπως έχουμε στην περίπτωση της Βυρμανίας ή στην Δημοκρατία της Κορέας, Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, είτε μέσω θεματικών ειδικών εντολών. Όπως πιστεύουμε ότι θα συμβεί για την ε, λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Και φυσικά θα πρέπει να εξασφαλιστεί μια συνέχεια σε διεθνές επίπεδο και μια συνέχεια για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αν θέλουμε να εξασφαλίσει την αξιοπιστία του. Ένα από τα σημεία της ημερήσιας διάταξης των ε, διαδοχικών συνόδων του Συμβουλίου είναι κάτι που θα μας απασχολήσει αργότερα σε επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης όταν θα εξετάσουμε την έκθεση Goldstone και την ειδική κατάσταση στη Γάζα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως σας πούμε και αργότερα, πιστεύει ότι η έκθεση Goldstone είναι πολύ σημαντική και σοβαρή και θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες και σοβαρές έρευνες για τις πιθανές παραβιάσεις ε, του διεθνούς δικαίου σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε θέματα διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Θα ήθελα τέλος να αναφερθώ στο πρόβλημα της αναθεώρησης του Συμβουλίου. Αυτή η χρονιά θα είναι κρίσιμη για τις διαπραγματεύσεις ως προς την αναθεώρηση της αξίας αυτού του Συμβουλίου που θα γίνει το 2011 η αναθεώρηση του έργου του Συμβουλίου. Ήδη ξεκινούν αυτές οι διαβουλεύσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να καταλήξει σε μια σαφή, συγκροτημένη και αποκρισταλωμένη στρατηγική ώστε να εθετήσουμε μια θέση που θα μας επιτρέπει να έχουμε και ενεργό συμμετοχή και να διατρανώσουμε τη δέσμευσή μας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και σίγουρα θα συνεχίσουμε ε, όπως κάναμε ανέκαθεν, να στηρίζουμε την ανεξαρτησία της ΥΠΑ της Αρμοστίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΙΕ, την ανεξαρτησία των ειδικών διαδικασιών, τη συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τη δυνατότητα του Συμβουλίου να αντιμετωπίσει κατάφορες σοβαρότητες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την θέσπιση εντολών αναχώρα. Η Ισπανική Προεδρία έχει επίγνωση ότι ανέλαβε την εκπεριτροπή Προεδρία σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα Ηνωμένα Έθνη και για το Συμβούλιο αυτό, προκειμένου να προωθήσει και να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο. Από αυτή την άποψη και η συνθήκη τη Λισαβόνα εγκαινιάζει μια νέα φάση. Μια νέα φάση για τι εξωτερικέ δράσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ευελπιστούμε ότι χάρη στη συνεργασία που θα γίνει υπό την αιγίδα της, είπα, της εκπροσώπου θα καταστήσει πιο ορατή και πιο στεντόρια τη φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα πλαίσια των εργασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θέλουμε ένα διαφανές, ενεργό Συμβούλιο που θα εκμεταλλευτεί αυτή τη μεταβατική φάση που διανύει η Ένωση με μια Προεδρία, την Ισπανική, που θα κάνει ό,τι μπορεί για να προλιάνει αυτό το έδαφος και θα υλοποιήσει το στόχο της προώθησης και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Να καλωσορίσουμε και στην πρώτη της παρουσία στην Ολομέλεια, πιστεύω, την Επίτροπο την κυρία Γεωργίεβα. Καλώς ήρθατε. Ε, και ελπίζουμε να έχετε μια εξαιρετική θητεία. Το λόγο λοιπόν τώρα εξ ονόματος της Επιτροπής η κυρία Γεωργίεβα. ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την θερμή αυτή υποδοχή και θεωρώ ότι είναι πολύ συμβολικό το ότι βρίσκομαι εδώ σήμερα για πρώτη φορά στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το οποίο εντάσσεται τόσο πολύ στο χαρτοφυλάκι των προτεραιοτήτων μου. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί απόλυτα με την παρουσίαση της Ισπανικής Προεδρίας. Θα ήθελα να προσθέσω δύο παρατηρήσεις σε αυτά που ήδη υπόθηκαν αναφορικά με τις προτεραιότητες και το πώς θα αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις προτεραιότητες αυτές. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τα κλιματικά ζητήματα, η, Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής ε, καταρτίζουν ε, ένα σχέδιο ψηφίσματος για τα δικαιώματα του παιδιού με ειδική στην καταπολέμηση της ε, σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών σε περιπτώσεις κρίσης και συγκρούσεων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας, τα παιδιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να διασφαλίσει ότι όλα αυτά τα θέματα θα τύχουν σωστή αντιμετώπιση στο ψήφισμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης θα συμμετάσχει σε ένα πάνελ για τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία και υπάρχει σε σύνδεση με τις εταιρικές μας πολιτικές καθώς ε, θα προσυπογράψουμε σύντομα τη Συμφωνία Ιων για τα άτομα με αναπηρία. Ένας άλλος τομέας ιδιαίτερο ενδιαφέροντος είναι το δικαίωμα στην τροφή που συνάδει με την ε, επίτευξη των στόχων της χιλιετίας καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα των ιστορικών εκτοπιστέντων που δεν προστατεύονται επαρκώς από διεθνείς συμβάσεις σε αντίθεση με τους πρόσφυγες. Δεύτερη παρατηρήση. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έγκριση από την Ολομέλεια των ε, καθολικών πρεδικών ε, εκθέσεων που πέρασαν από τη ε, διαδικασία αυτή το Δεκέμβριο. Είναι πολύ σημαντική στιγμή αυτή, κατά την οποία τα κράτη και οι αναθεωρήσεις τους μπορούν να δημοσιεύσουν τις παρατηρήσεις τους για την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Εκ παραλλήλου, τα κράτη μπορεί να επιλέξουν να ζητήσουν διεθνή αρρωγή για την εφαρμογή των δεσμεύσεων αυτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει ανοιχτή για τις συζητήσεις με τους εταίρους προκειμένου να ε, υποστηρίξει την εφαρμογή των ε, εκθέσεων αυτών. Επίσης, όπως είπε η Ισπανική Προεδρία, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο αντίκτυπος της διαδικασίας αυτής εξαρτάται καταρχάς από την διαφάνεια και τον ανοιχτό χαρακτήρα που επιδεικνύουν τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Γιατί μπορεί να είμαστε αποτελεσματικοί μόνο αν θέσουμε εμείς το σωστό παράδειγμα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα περνάμε στους ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Πρώτη είναι η κυρία ε, για δύο λεπτά. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπέ, κύριε Προεδρεύοντα. Καλωσορίζω το γεγονός ότι θα εγκρίνει ε, το Κοινοβούλιο το σχετικό ψήφισμα για το Συμβούλιο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Επίσης, καλωσορίζω το γεγονό ότι θα αποστείλουμε ε, ε, αποστολή στο Συμβούλιο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων από τις συστάσεις μας προς το Συμβούλιο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων αναφέρω πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η σύνοδος και η πιο σημαντική που θα λάβει η χώρα το 2010 και σε όλες τις επαφές της υψηλού επίπεδου έχουν αναφερθεί ήδη πολλά σημαντικά θέματα από τον Υπουργό και από την Επίτροπο, όπως για παράδειγμα ο αντίκτυπος της χρηματοοικονομικής κρίσης στην κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Καλωσορίζουμε το γεγονός ότι οι Αμερικάνοι ομολογοί μας ε, δεσμεύονται σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Ωστόσο, κάποιες χώρες προσπαθούν να υποσκάψουν την αξιοπιστία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το Ιράν έχει ε, υποδείξει, ανέφερε ότι μπορεί να ζητήσει να εκλεχθεί στο Συμβουλίο. Θα ήταν πάρα πολύ λυπηρό αυτό, γιατί αυτό θα αύξανε τον αριθμό χωρών με προβληματική κατάσταση και ιστορικό σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και το Συμβούλιο των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων θα κινδύνευε να καταστεί εξίσου αναποτελεσματικό όπως και το προηγούμενο Συμβούλιο και άρα διακυβεύεται η όλη αξιοπιστία του Συμβουλίου και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να διατηρήσουμε το κύρος του Συμβουλίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να, να καλωσορίσω τις ε, προτεραιότητες του Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων γιατί ζητήσαμε στη, στον ΟΗΕ να αυξηθεί η δέσμευση του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και επίσης συνεργαζόμαστε με τρίτες χώρες ως ε, τμήμα των κοινών προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και χαίρομαι που στην ε, Γενέβη ανακοινώθηκε, θα ανακοινωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωταθλητή σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πρωταθλητέ και στα πλαίσια του Συμβουλίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, γιατί παραμένει υπερβολικά υψηλό ο πολιτικό χαρακτήρα ε, του Συμβουλίου. Για παράδειγμα, θα ζητηθεί λόγος, ε, ο λόγος για να υποστηριχθεί η θέση της Σρι σε ό,τι αφορά το ιστορικό της τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις καταχρήσεις. Στο Κοινοβούλιο αυτό συμφωνούμε με πολλές από τις αρχές που είναι η Ισπανική Προεδρία σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα ήθελα να συμφωνήσω με την κυρία Ανδροκίν ότι θα είναι πραγματικά, θα σημαίνει το θάνατο του Συμβουλίου αν εκλεχθεί ε, χωρίς αντίρρηση το Ιράν όπως φοβούνται ορισμένοι. Το πιο, η πιο ισχυρή δοκιμασία για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι το πώς αντιμετωπίζουμε τις καταχρήσεις. Και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα, χαίρομαι που οι Ηνωμένε Πολιτείε και όλες οι οργανώσεις που συναντήθηκαν το Φεβρουάριο μίλησαν κατά της ε, μυστικής κράτησης ε, των ατόμων. Πάντα θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί την κριτική εφόσον περιμένουμε και οι ομολογή μας να κάνουν το ίδιο. Η κυρία Ότζουλαντ για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, εμείς οι φιλελεύθεροι Θέλουμε να είναι ορατή η Ευρωπαϊκή Ένωση στην, στα εγγένεια της 13ης Συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό ε, του ψηφίσματος. Ήθελα να επισημάνω τις παραγράφους 9 και 13 για το Ιράν. Για μας τους φιλελευθέρους είναι απαράδεκτο το ότι το Συμβούλιο δεν μπορεί, για να μην σας πω ότι δεν θέλει, να αντιδράσει με την δέουσα ταχύτητα όσον αφορά αυτή την ανθρωπιστική κρίση σε Ουή, Νέα, Ιεμένη, Ιράν, Αφγανιστάν, Ιράκ γιατί το Συμβούλιο των Δικαιωμάτων είναι ένας φορέας που όλες οι αναγνωμένες χώρες της εκπροσωπεί. Έχει παρακολουθήσει την κατάσταση στην ανθρωπίνη δικαιώματα σε αυτές τις χώρες. Σε όλα τα κράτη-μέλη. η βραδύτητα αντίδραση του Συμβουλίου δείχνει την αδυναμία του φορέα αυτού. Δείχνει την αδυναμία του να κληρώσει τα καθήκοντά του. Είναι μια αδυναμία η οποία φάνηκε και από την υποψηφιότητα. Τι έγινε το Μάιο τόσο πάντων εκλογέ. Είναι παράλογη αυτή η κατάσταση. Είναι υποψήφιοι για να μπουν στο Συμβούλιο Θεωρημένων Δικαιωμάτων. Είναι κράτος καταστολής και καταπίεσης με μηχανισμούς αντίστοιχους. Είναι θρησκευτικό κράτος. Θα ήθελα ο ύποδος εκπρόσωπος να υιοθετήσει κάποια θέση πάρα πολύ σκληρή και έτσι να ασκήσει πίεση στη χώρα αυτή. Ε, Σας ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εδώ μια καταπληκτική ευκαιρία ούτως ώστε να αναβαθμίσει την ευαισθησία της, ε, ε, της διεθνούς κοινότητας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα έτσι και έτσι μπορεί κάτι να κάνει το Συμβούλιο και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να προωθήσει την ε, έκθεση Γκόλστον για την Γάζα και έτσι να αντιδράσει όσον αφορά αυτές τις ε, παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επομένω, και εμεί θέλουμε να μα πει πάντω εκπρόσωπο ακριβώ πώ έχει η κατάσταση. Ακριβώ τι κάνει, τι πρεσβεύει το κάθε κράτο μέλο σε σχέση με αυτή την τόσο σημαντική έκθεση. Και έτσι να εξασφαλιστεί ότι τηρείται το διεθνέ δίκαιο και προσάγονται ενώπιον των δικαστηρίων αυτοί που παρεμβαίνουν ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει όλα αυτά τα ακριβή θέματα να επιληθούν. Θα πρέπει να καταλάβει ποιο την προσπάθεια η Ευρώπη και έτσι να καταπολεμήσει τέτοιου είδου πράξει. Κάτι να γίνει για αυτού που είναι φυλακισμένοι, για αυτού που υποφέρουν και θα πρέπει μένουν στα κράτη-μέλη να κάτσουν και να σκεφτούν Μήπω τα ίδια έχουν παραβιάσει τα ανθρωπινά δικαιώματα ή στο παρελθόν. Δεν είναι εδώ να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Να, επομένω, πώ μα δίνει τώρα μια ευκαιρία να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε και το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο. Ούτω ώστε να υιοθετήσουμε μια δυναμική στάση και έτσι να μπορούμε να προβάλλουμε το μήνυμα. Πρόεδρε, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το ΟΗΕ αναμφίβολα έχει ιδιαίτερα ε, θετικούς στόχους, αλλά πολλές ε, χώρες ε, υπονομεύουν αυτό το ρόλο όπως η Κούβα, οι άλλες χώρες όπως το Ιράν που είναι υποψήφιο για μέλος. Θα πρέπει λοιπόν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει σε επαφή με το επίπεδο του ΟΗΕ. Γίνονται κάποιες καλές προσπάθειες όσον αφορά την προστασία των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα των παιδιών, όμως πολλές φορές διαφεύγουν του δημοκρατικού ελέγχου. Εδώ το ψήφισμά μας τονίζει ότι η 13η Σύνοδος ε, δεν καταφέρνει να υπογραμμίσει τα προβλήματα που υπάρχουν στη Γινεγουινέα Κόνακρη, στην Ιεμένη, στο Ιράν, στο Αφγανιστάν. Επίσης για το θέμα της CIA και των εκτάκτων ε, επιστροφών ε, ε, διαμετακομίσεων φυλακισμένων θα πρέπει να το σκεφτούμε δύο φορές πριν να επιτεθούμε κατά των Αμερικανών συμμάχων μας. Mr. Chairman, Κύριε Πρόεδρε, ενώ η Κομισιόν θέλει να υποστηρίξει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμεί πιστεύουμε ότι ο 20 ο αιώνας ε, δεν έχει προχωρήσει και πάρα πολύ. Ε, η, Ευρωπα... η Κομισιόν θεωρεί πω είναι παγκόσμιο παίκτη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φαίνεται να είναι έτοιμη να κρίνει του άλλου και να προσφέρει βοήθεια και συμβουλή. Ωστόσο θα πρέπει να κάνει λίγη αυτοκριτική. Θεωρώ πω είναι εξαιρετικά ηρωνικό ότι ενώ εμεί υποστηρίζουμε τα δικαιώματα των ε, πολιτών του Κασμίρ και του υποστηρίζουμε στην αυτοδιάθεση, πράγμα το οποίο του υποσχέθηκε προσχέθηκε το 1947 ο ΙΕ, η Κομισιόν από την άλλη πλευρά ενεργά προσπαθεί να αφαιρέσει αρμοδιότητε από τα ίδια τη τα κράτη-μέλη σε τομεί ε, πολιτική που ενθαρρύνονται και από την ε, συνθήκη τη Λισαβόνα. Και αυτό με φέρνει στο θέμα του δημοψηφίσματο που ε, ήταν υπόσχεση προ το Βρετανικό εκλογικό σώμα και ποτέ δεν συνέβη. Γι' αυτό κύριε Πρόεδρε το δικό μου εκλογικό σώμα περιμένει την αυτοδιάθεση μαζί με του πολίτε του Κασμίρ. Ευχαριστώ. Κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω πως είναι μια ονειρεμένη ευκαιρία για να επιβεβαιώσουμε την ε, καθολικότητα και την ε, ε, γενική ισχύ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ συχνά έχουμε την ευκαιρία να το δηλώσουμε, όπω στην έκθεση Χαβιέρ για τα εγκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και με διάφορα ψηφίσματα, όπω πρόσφατα το κάνουμε με το Ιράν. Άλλοι συνάδελφοι στι παρεμβάσει του ε, εκτίμησαν πω ήταν παράδοξο ορισμένε χώρε που έχουν πραγματικά πολύ κακό ρεκόρ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα αναλαμβάνουν να επιβλέπουν την τήρηση αυτών των ίδιων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να συμμετέχουν σε όργανο το ΟΗΕ. Εγώ πιστεύω πως αυτά τα όργανα, αυτό το Συμβούλιο πραγματικά θα ήταν τελείως άχρηστο αν δεν έχει πλέον την ηθική, το ηθικό κύρος που του να το επιτρέπει να όντως να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, Πρόεδρε, να σας θυμίσω πως αυτές τις μέρες, αυτή την εβδομάδα, μιλήσαμε για την έκδοση από την Κούβα ενός συναδέλφου της, ε, του σώματός μας. Εγώ θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου για το θάνατο ενός 52χρονου ε, οικοδόμου που πέθανε μετά από απεργία πείνας, μετά από μακρά ε, απάνθρωπη κράτηση ο κύριος Λιζάρντο Σάντσες που, που είναι πολύ κοντά στην ε, σοσιαλδημοκρατία στην Κούβα είπε πως αυτός ο θάνατος μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Θεωρεί πως αυτός ο θάνατος είναι μια δολοφονία υπό νομική κάλυψη. Ξέρουμε βέβαια ήδη τη θέση του Προεδρεύοντος του Συμβουλίου. Εγώ σας ρωτώ κύριε Επίτροπε αν πιστεύετε πως μέσα σε μια ηθική και δημοκρατική ε, θέση θεωρείται ότι απέναντι σε ένα τόσο αξιοθρύνητο γεγονό όπω ο θάνατο του κυρίου Ζαπάντα είναι προβλέψιμο ε, και προβλεπταίο το να βελτιώσουμε τι σχέσει μα με την Κούβα σε υψηλότερο επίπεδο. Θα Καλωσορίσω στην αίθουσα τον μακαριότατο του Αρχιεπίσκοπο Χόρχε Ορτίγα, του συνοδεύοντε αυτών επισκόπου και ολόκληρη την αντιπροσωπεία τη Επισκοπική Διάσκεψη τη Πορτογαλία. Είστε εδώ. Καλώς ήρθατε. Μακαριότατε. Δράτω με τις ευκαιρίες. Δράτω με τις ευκαιρίες για να εκφράσω την αλληλεγγύη μας και τα συλληπιτήριά μας στο λαό της Πορτογαλίας και ειδικότερα στο λαό της Μαδέρα που δοκιμάστηκαν τόσο σκληρά τις τελευταίες αυτές ημέρες. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας τους συνοδεύουν.